Allora, riprendiamo, cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Πάμε σε επεξηγήσει ψήφων. Ελέσσα για την απαλλαγή 2017, Γενικό υπολογισμό. Συνάδελφε πεισίλε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. στήριξε αυτή την έκθεση για την απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Τσέχος λυπάμαι που ένα μεγάλο τμήμα της έκθεσης ασχολεί, ασχολείται με τον κύριο Μπάμπης, τον Πρωθυπουργό μας. Γιατί στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίε τώρα τυπικά δεν είναι δικέ του. Πρόκειται όμω ουσιαστικά για κατάχρηση πόρων, ευρωπαϊκών πόρων. Η δικαστική εξέταση είναι να εξελίξει και θα πρέπει να περιμένουμε σε, για να δούμε σε τι βαθμό οι ενέργειες του κ. Μπάμπης παραβιάζουν τον νόμο. Θα πρέπει να περιμένουμε γι' αυτό. Ο κύριος... Συνάδελφε Άναν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, για τα λεφτά πάντα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πολύ καλός μηχανισμός για να παίρνει λεφτά από τους φορολογούμενους και να τα αναδιανέμει στους τυχερούς. Αυτοί που είναι δηλαδή άμεσα ή έμεσα τμήμα του συστήματος. Βέβαια δεν είναι η μόνη. Κάθε σύστημα διακυβέρνησης έχει και αυτή την πλευρά. Αλλά αυτό που είναι μοναδικό είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο αυτές τις ε, ε, παράνομες ενέργειες τελειοποιεί όλο και περισσότερο αυτή την κακή πλευρά. Ε, οποιαδήποτε νομοθετική συνέλευση θέλει οπωσδήποτε να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Αλλά για το καλό της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, το Κοινοβούλιο τελικά πάντα συντάσσεται με την Επιτροπή στο όνομα της περισσότερης συνοποίησης. Και αυτό ήταν το πρόβλημα από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Έκθεση του Γενικού Προπολογισμού για το δικαστήριο. Ο κύριος μέσας παρακαλώ, ένα λεπτό. <clears throat> Δεν είναι παρόν. <clears throat> Δεν είναι παρόν. Καλώς. Λοιπόν, επόμενη έκθεση. Σαρβαμά. Απαγωγή, ε, συγγνώμη, απαλλαγή 2017, Μάιερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα 500 εκατομμύρια που θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή, ε, ο Ευρωπαϊκός Φορέας ε, Φαρμάκων γιατί δεν μπορεί να βγει από το συμβόλιο που είχε στο, για τα γραφεία του στο Λονδίνο είναι τρομερή απώλεια. Και έτσι θα χάσουμε πόρου για το προσωπικό και για έρευνα. Και είναι πολύ ψηλού επίπεδου αυτός ο οργανισμό στι τελευταίε δύο δεκαετίες έχει παίξει ανεκτήμητο ρόλο. Απλοποιεί και προωθεί του κανόνε για τα φάρμακα και επιτρέπει να εγκριθούν σε όλα τα κράτη-μέλη με τη μία ε, τα φάρμακα. Αλλά δυστυχώ αυτό δεν θα ισχύει πλέον για τη χώρα μου. Και ήδη στην εκλογική μου περιφέρεια ένας ε, φαρμακοβιομήχανος δημιούργησε ένα παράλληλο μηχανισμό ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να, πολλά, να πωλεί τα προϊόντα του και στην Ένωση. Αυτό σημαίνει περισσότερο κόστος και λιγότερα χρήματα για την και ανάπτυξη και αυτό σημαίνει ότι η Βρετανία θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα για τα φαρμακά τη. Και θα έχουμε λιγότερα χρήματα λοιπόν για τι άλλε δαπάνε ε, του συστήματο υγεία. Είναι το αντίθετο ακριβώ αυτό, από αυτό που πίστευαν ότι ψήφισαν όσοι ψήφισαν υπέρ του Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Σαρβαμά και πάλι ο κύριος μη τον οποίον δεν βλέπω ούτε τώρα, είναι στην αίθουσα. Όχι. Οπότε, επόμενη έκθεση. Παντζέρι, Πρέντα, Έγγελ, Γκέρενς. Ο κύριος Τάνοκ, δύο λεπτά παρακαλώ, από πλευρά της ομάδας του. Κύριε Πρόεδρε, από πλευρά τη ομάδα μου θέλω να ευχαριστήσω του συνεισηγητέ και του ε, άλλου κοιόδη για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο ε, συμφωνήσαμε επί συμβαστικού κειμένου για αυτό το πολύ ευρύ και δύσκολο θέμα. Χαιρετώ, χαιρετίζω το γεγονό ότι έχουμε ένα ενιοποιημένο μέσο, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έτσι θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και θα αξιοποιήσουμε καλύτερα του πόρου τους πόρους μα ε, στου τομεί αυτού. Τώρα που <clears throat> η μετάβαση η, ε, δημιουργεί προβλήματα στις χώρες του Νότου λόγω και της παρέμβασης ε, της Ρωσίας η πολιτική γειτονία είναι πρωτής της σημασίας. Προσωπικά Καλωσορίζω αυτό το πλήρως ενοποιημένο μέσο. Ξέρω ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες και στην αίθουσα και στην ομάδα μου για ορισμένε πλευρέ του. Και αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει τώρα να συνεχιστούν κατά την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. <clears throat> Επειδή υπάρχει πολύ αυστηρός γεωγραφικός περιορισμός του μέσου, δεν θεωρώ ότι ε, θα επιβαρυνθούν ορισμένα τμήματα της γειτονίας εις βάρος άλλων θα προτιμηθούν εις βάρος άλλων. Και το γεγονό ότι το 95% τη χρηματοδότηση θα ε, είναι με βάση τα κριτήρια του ΟΣΑ πρέπει να μας καθησυχάζει. Είναι σοβαρή αύξηση με βάση το 92% που είχε προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζω και την ε, δημιουργία ενός πολύ πιο φιλόδοξου σύν Οι αλλαγές αυτές θα αλλάξουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, τράπεζα Επενδύσεων. Και Χαίρομαι που ένα ελάχιστο ποσοστό χρηματοδοτήσεων θα δίδεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπως ε, προβλέπει το, η τροπολογία 52. Λυπάμαι που δεν θα είμαι εδώ για τι τελικέ διαπραγματεύσει για το μέσο αυτό στην επόμενη θεία και λυπάμαι που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει σε ένα εγχείρημα που υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη με τις διαστάσεις της ε, μπορεί να παίξει το ρόλο της αν όλοι συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έκθεση Σαλαφράνκα Φλέκερστάιν. Συνάδελφε Ντανζό, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει μέρος του προπολογισμού της στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη χωρών που είναι στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια για παράδειγμα. Απόλυτα θέμητο αυτό. Η γαλλική αντιπροσωπεία όμως κράτησε θέση αποχής για την έκθεση αυτή για να εκφράσει τις επιφυλάξεις της σε δύο σημεία της πρότασης αυτής, η πατρία. Πρώτα απ' όλα, οι πόροι, τα κονδύλια που πηγαίνουν στην Τουρκία, που είναι μία μη ευρωπαϊκή χώρα, πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικά ε, μεγάλα για να στηρίξουμε την ε, μετανάστευση. Από την άλλη μεριά, έτσι όπως ονομάζεται αυτός ο προϋπολογισμός, που είναι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, ε, δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις οι οποίες μας ζημιώνουν δεν συμφωνούμε όλοι. Δεν πρόκειται για μια ε, διαδικασία που είναι αυτόματη. Κάποιοι από τους δικαιούχους των πρωτοξιακών κονδυλίων δεν είναι καν υποψήφιες χώρες. Θα ήταν καλύτερο να σταθμίσουμε διαφορετικά το μηχανισμό αυτόν και να τον αποσυνδέσουμε πλήρως από την λογική της διεύρυνσης. Ευχαριστώ, ήταν τελευταία παρέμβαση. Οπότε διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3. Σας εύχομαι λοιπόν καλή όρεξη.